οποιοδήποτε σενάριο. Δεν θα πρέπει να ε, προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε όλες τις ε, τριβές ε, στα σύνορα χωρίς το επίμαχο θέμα του backstop. Νομίζω αυτή ήταν η απάντηση πάντοτε και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητέ Μισολμπάνια συνάδελφοι. Νομίζουμε ότι από τη συζήτηση καθίσταται σαφές, όπως και από πολλές πρωτεύουσε, ότι υπάρχει ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27 κράτη-μέλη έχουν την ίδια αντίληψη. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει ενότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς θα εμείνουμε στην ενότητά μας και στην ε, ε, ακαιρεότητα της ε, ενιαία αγορά. Το δεύτερο, χθες υπήρξε μια συμμαχία ε, των αρνητών. Από τη μία είναι οι σκληροί αποχωρητέ, από την άλλη είναι αυτοί που θέλουν να παραμείνουν και συμφωνούν σε αυτό που δεν θέλουν. Η Τερίζα Μέη προσπάθησε να προσφέρει μια ε, επικοδομητική λύση. Τώρα όμως λέει ότι θα μιλήσει με την αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχει μιλήσει από δύο χρόνια θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια επικοδομητική λύση από το Βρετανικό Κοινοβούλιο τελικά επί της οποίας να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ο κύριος Κόρμπιν είπε ότι θέλει η Τελωνιακή Ένωση. Ε, ας κάνει αυτή την πρόταση. Ας βρει πλειοψηφία για αυτήν. Δεν θα είχαμε πρόβλημα. Και θα μας επέτρεπε να βρούμε μια λύση. Θα ήταν πολύ καλό κάτι τέτοιο. Αν υπάρξει μια επικοδομητική λύση, Βεβαίω, να την εγκρίνουμε. Πέρασε τώρα η εποχή που θα έπρεπε οι κομματικές και προσωπικές φιλοδοξίες να αποτρέπουν την εξέβρεση λύσης. Πρέπει λοιπόν να τολμήσουν οι Βρετανοί να έχουν αυτό το θάρρος. Ο κύριος Βάιντενχολτσερ. Ευχαριστώ. Είναι ιστορική στιγμή. Όπως ξέρουμε η ιστορία πάντα μας εκπλήσει. Όταν ξεκινήσαμε τη θητεία μας το 2015, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα κάναμε σήμερα μια τέτοια συζήτηση. Ούτε καν το 2016, όταν συζητούσαμε το απροσδόκητο αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος. Πέρασαν έκτοτε 900 μέρες μέχρι να λάβει μια απόφαση που να έχει έννοια το Βρετανικό Κοινοβούλιο περάσαμε μήνες αβεβαιότητας και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Το μέλλον εξακολουθεί να είναι απρόβλεπτο. Απόλυτα σκοτεινό. Ένα όμως είναι σαφές. Τελειώνει ο χρόνος. Θα λήξει ο χρόνος. Σε 70 μέρες υπάρχει κίνδυνος να υπνοβατήσει αυτό το μεγάλο έθνος προς την καταστροφή. Θα πρέπει να καταλάβετε ως καμπανάκι αυτά που έγιναν χθε. Θα πρέπει να συζητήσουμε τη λογοδοσία ε, των κυβερνητών. Πώς είναι δυνατόν μια μικρή ελίτ για κοντόθωρους λόγους να έχει όμοιρο ολόκληρη τη χώρα. Είναι σαφές ότι απέτυχαν οι Βρετανοί συντηρητικοί. Αλλά τώρα το θέμα δεν είναι να επιμένουμε ποιος έχει δίκιο, ούτε να επιχειρήσει κανείς να εκδικηθεί ή να επιβάλλει αντίπεινα. Πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα προς το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. Οι απλοί άνθρωποι στη Βρετανία έχουν πολλά να χάσουν εάν υπάρξει σκληρή αποχώρηση. Εμείς, τα 27 κράτη-μέλη που μείναμε ενωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο και για να υπάρξουν πραγματιστικές λύσεις να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημίες. μπορείτε να βασιστείτε στην ομάδα τη δική μας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τα τελευταία 40 χρόνια δεν ξεχνάμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμβάλει τρομερά στο κοινό μα εγχείρημα θα μας λείψει η εμπειρογνωμοσύνη των Βρετανών συναδέλφων μας. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αποτελέσματα στην προσπάθειά μας. Θέλουμε λοιπόν βεβαιότητα για το τι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε σαφή μηνύματα. Θα μπορούσε μια νέα ψηφοφορία να μας δώσει αυτό το αποτέλεσμα, ένα νέο ψήφισμα. Ο, Βρετανός, ο Βρετανικός λαός θα έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του και κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ε, δεν ξέρει γιατί ψηφίζει ο ψηφοφόρος. Δεν θέλω να παρέμβω στα εσωτερικά σας, αλλά θα καλοδεχόμεθα οποιαδήποτε απόφαση να παραμείνετε. Στείλαμε μία επιστολή μαζί με 40 συναδέλφους αυτή τη εβδομάδα για να καταστεί σαφές ότι θέλουμε να μείνετε και θα σας καλωσορίσουμε με ανοιχτές αγκάλες εάν επανέλθετε. Κύριε Βάντεν Χόλτσερ, υπάρχει μια μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε. Όχι, ευχαριστώ. Σμιθ. Σας κατανοώ. Έχετε όλοι να αντιμετωπίσετε αυτές τις αχλαμάρες. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά παρατηρήσατε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι και τόσο ενωμένο και με την συντηρητική κυβέρνηση δυστυχώς έχει διαιρεθεί ε, ακόμα περισσότερο. Και εγώ εκπροσωπώ τη σκοτία ε, και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στην Ηνωμένη Ευρώπη, θέλουμε να μείνουμε στην οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών. Αλλά έχετε να αντιμετωπίσετε το Ηνωμένο Βασίλειο ως έχει πρέπει να σεβαστείτε τη συνταγματική τάξη της συγκεκριμένη χώρας. Η θέση της Σκοτίας είναι σαφής. Δεν υπάρχει καλό Brexit. Είναι κακό για τη Σκοτία, κακό για το Ηνωμένο Βασίλειο, κακό για την Ενωμένη Ευρώπη. Η προσπάθειά μου δεν είναι να μετριάσω τις αρνητικές συνέπειες του Brexit, αλλά να σταματήσω τον Brexit. Και υπάρχουν πολλοί Βρετανοί οι οποίοι ανήκουν σε πολλά κόμματα συνάδελφοι που προσπαθούν να βρουν κάποια λογική λύση. Πρώτον, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα θέλετε να παραμείνουμε, θέλουμε χρόνο. Και ίσως να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη διαδικασία αυτή μόνο αν συνεργαστούμε στενά και τότε ίσως η κυβέρνηση της, του Ηνωμένου Βασιλείου ακούσει και άλλες φωνές και όχι μόνο τις δικές της. Πάρα πολλοί πολίτες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου αγχώνονται οι Βρετανοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ευθύνε για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα αυτά, να διευκρινίσουμε την κατάστασή τους, να τους διασφαλίσουμε το μέλλον τους ε, και να μην τους δώσουμε την δυνατότητα να παραμείνουν μέσα σε μια διαδικασία την οποία δεν ελέγχουν. Είναι καθήκον προς τους πολίτες μας. Η Επιτροπή έκανε προσπάθειες για να υπάρξει εγγύηση για τα δικαιώματα αυτά, αλλά λόγω της απουσίας δράσης από πλευρά της Βρετανικής κυβέρνησης πρέπει εμείς να αναλάβουμε δράση. Νομίζω ότι αυτά τα δύο, ε, οι δύο στόχοι αυτοί μπορεί ε, να βοηθήσουν. Θα πρέπει έτσι να βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί το Westminster. Έχετε μία μπλε κάρτα, θέλετε να απαντήσετε. Από ποιον είναι η μπλε κάρτα, λέει ο κ. Σμιτ. Όχι, όχι, δεν θα δώσω περισσότερο οξυγόνο στον Κόμπερν από ήδη καταναλώνει. Η κυρία Σπινέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προοπτική μια έλλειψη συμφωνία για το Brexit αντιπροσωπεύει ένα, μια σοβαρή βλάβη για τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής πάνω στην οποία οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδία κάποτε θα κληθούν να αποφασίσουν, αλλά και για τους Βρετανούς πολίτες που ζουν ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ορίζοντας είναι σκοτεινός. Η απουσία μιας συμφωνίας θα του στερήσει τα δικαιώματα ελευθερίας διακίνησης. Από τη σημερινή εκκρεμότητα θα περάσουν στη νομική αβεβαιότητα, σε ένα εφιάλτη. Είναι δύσκολο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την τεράστια σύγχυση την οποία έχει δημιουργήσει η εκτελεστική εξουσία αν δεν εκφραστεί για μια ακόμη φορά ο λαός. Αν επιβεβαιωθεί το no deal, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας να ευθυγραμμιστούν οι εθνικές πρακτικές στα λεγόμενα best practice και δίδοντας εγγυήσεις στους Βρετανούς πολίτες για την ελεύθερη διακίνησή τους. Ακόμα πιο σοβαρή είναι η θέση των τριών εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο που κινδυνεύουν να βρεθούν και αυτοί θύματα του εχθρικού περιβάλλοντος που προωθούν οι συντηρητικοί από το 2012 οι υποσχέσεις της ΜΕΙ μπορεί να αναιρεθούν με μια σύντομη ψηφοφορία από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Μόνο αν εφαρμοστούν οι προβλέψεις της συμφωνίας θα τους δώσει μια νομική ασφάλεια. Η προστασία νομική των δικαιωμάτων αυτών είναι δυνατή εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύσει μονομερώς τους πολίτες της Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη και οδηγηθούμε εκ νέου σε μια προκαταρκτική συμφωνία Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου που προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κεφάλαιο για τα δικαιώματα. Αυτό είναι κρίσιμο, αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ και το επαναλαμβάνω αυτό στον κύριο Μπαρνιέ Η κυρία Άτκινσον έχει το λόγο. Δεν είμαστε λίγο ε, απογοητευμένοι σήμερα. Κυρία Μέη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ιούνκερ, τον κύριο Φερχόφσταντ, ε, ε, οι οποίοι, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω του όσοι ψήφισαν 17 εκατομμύρια, οι οποίοι ψήφισαν για το Brexit και να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε GPOC, δεν είμαστε θηγατρικοί ε, των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρξε προδοσία. Έχουμε Έχουμε μια κυβέρνηση, μια πρωθυπουργό και αντιπολίτευση 17,2 εκατομμύρια που ε, ψήφισαν ε, ή ψήφισαν μαζί με με, τους, με αυτούς των Ηνωμένων Πολιτειών του Commonwealth. Μπορούμε ε, να ακολουθήσουμε τους κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού ε, Εμπορία. Και έχουμε του 17,4 εκατομμύρια που ψήφισαν για το Brexit. Θα κάνουμε και πάλι τη Μεγάλη Βρετανία μεγάλη. Θα ήθελα να ξαναγίνει μεγάλη η Μεγάλη Βρετανία και πάλι στον μεγάλο ευρύτερο κόσμο. Επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά, ε, η κυρία Κέλλη. Ναι, ε, συμφωνώ με τα περισσότερα πράγματα που λέχθηκαν εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι η ψηφοφορία εχθές το βράδυ ήταν κάτι το προβλέψιμο και οφείλω να ομολογήσω ότι η ενότητα των 27 είναι θαυμαστή χάρη στο Μισελ Μπαρνιέ ε, στην εργασία του και στην εργασία όσων συμμετείχαν σε αυτό το έργο. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σχόλιο που λέχθηκε ε, χτες το να προσπαθήσει να πει κανείς αυτό σε αυτούς που ε, έχουν αυτά τα σύνορα που προστατεύονται από τους Βρετανούς ε, στρατιώτες το να πει κανείς ότι αυτά όλα δεν είναι χρήσιμα και χάρη σε βία που υπήρξε είχαμε τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και να πούμε ότι ο, ο κύριος Μπαρνιέ και ε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάνανε το παν για να εξασφαλίσουν ότι θα προστατευτεί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και η ειρήνη σε όλη την Ιρλανδία θα ήθελα να πω στην συνάδελφο Άντερσον ότι δεν είναι η στιγμή ε, να ε, κάνουμε τέτοια έκκληση. Δεν είναι η θέση ε, της Ιρλανδικής κυβέρνησης του λαού της Ιρλανδίας παρόλο που ευχόμαστε μια ενωμένη Ιρλανδία. Δεν νομίζω ότι αυτό ήθελε ο πληθυσμός. Ο μεγάλος φόβος είναι να μην υπάρξει ε, συμφωνία. Το να βγει με τρόπο άτακτο από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση η Μεγάλη Βρετανία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτέλεσμα. Αλλά ο φόβος είναι η Μεγάλη Βρετανία να λάβει μια απόφαση που δεν είναι πράγματι αυτό ε, που θέλει, αυτό που θέλει ο λαός. Δεν θέλει ένα τέτοιο σενάριο. Θα πρέπει να μπορεί να εκφραστεί και θα πρέπει ότι το πιο ε, έξυπνο θα ήταν να ξανασυμβουλευτούμε αυτούς ψήφισαν ο Βρετανικός λαός. Είναι πραγματικά αυτό που ήθελε. Νομίζω ότι θα πει όχι αν ξαναερωτηθεί. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά στον κύριο Ευχαριστώ. Ας είμαστε σαφείς. Πώς καταλήξαμε εδώ. Ε, η κυβέρνηση ενδιαφερόταν μόνο για τα συμφέροντα του Συντηρητικού Κόμματο και δεν τα προστάτευσε ούτε καν πολύ καλά. Έτσι καταλήξαμε εδώ. Η κυβέρνηση αυτή αρκεί, θα έπρεπε να φύγει. Αλλά αυτή η συζήτηση φυσικά πρέπει να γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οποιοδήποτε κόμμα είναι στην εξουσία θα πρέπει να κάνει αυτή την επιλογή σε σχέση με τον Brexit. Ή θα αποχωρήσει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφοντας ε, θέσεις εργασίας, καταστρέφοντας το περιβάλλον, καταστρέφοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων ή παραμένεις εντός της Ένωσης και χάνεις οποιαδήποτε δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις δομές. Αυτή είναι η επιλογή εάν υπάρξει Brexit. Κανένα από αυτά τα δύο δεν είναι σωστά για καμία χώρα και σίγουρα όχι για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά εγώ θέλω να σα δώσω ένα μήνυμα ελπίδα για την Βρετανία. Χάρη σε αυτού του τύπου απέναντι που είναι τόσο περίεργοι, καταλήξαμε στο μεγαλύτερο φιλοευρωπαϊκό κίνημα στην Ήπειρο. Έχουμε εκατομμύρια πολιτών μα που είναι δεδεθμένοι να βγουν έξω για να περασπιστούν τι αξίε τη Ένωση και να πούνε ανοιχτά ότι είμαστε περήφανοι για αυτά που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά που θα επιτύχει. Θα υπερασπιστούμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Θα υπερασπιστούμε τι δομέ τη Ένωση. Όχι αυτέ που έχουμε τώρα, αλλά και αυτέ που θα αποκτήσει το μέλλον η Ένωση. Και αυτέ οι ανοησίε και ε, τα ψέματα που λένε, από την άλλη μεριά, καθιστούν σαφέ ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για άτακτη αποχώρηση. Εάν θα υπάρξουν νέε εκλογέ, εάν θα υπάρξει νέο δημοψήφισμα, εάν θα υπάρξει νέα πλειοψηφία για κάποια άλλη λύση, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Σα παρακαλούμε, συνάδελφοι, α μην αφήσετε τη διαδικασία να νικήσει την πολιτική. Έχουμε δυνατότητα να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία. Θέλουμε τη στήριξή σα και τη φιλία σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σκοτ Κέιτσο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είδα την ιστορική ψηφοφορία στο Westminster, εδώ στο Στρασβούργο με συναδέλφου ε, από όλε τι χώρε που ανησυχούν ιδιαίτερα για την κρίση αυτή. Πολλοί ελπίζουν να βρούμε έναν τρόπο να μείνουμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για τη στήριξή σας. Το Brexit είναι η ε, αποτυχία της ηγεσία. Απέτυχε η Τερίσα Μέη. Ε, ασχολήθηκε μόνο με τις ανάγκες του κομματός της. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν απέτυχε στο συνταγματικό δικαίωμά του, ε, συνταγματική υποχρέωσή του να αντισταθεί στο Brexit. Η χώρα μας λοιπόν είναι σε απόγνωση. Αλλά το Brexit είναι και έλλειψη αλληλεγγύης. Οι παλαιότερες γενιές αγνοούν τους πόθους των νέων. Πολλοί Βρετανοί ξέχασαν τους άλλους πολίτες που είναι στην κοινότητά μα και παίζουν ζωτικό ρόλο, ό, συναδέλφου, του τους ε, του, τους που ζουν εκτός ε, Βρετανίας. Πολλοί είδαν τη ζωή τους να αντιστρέφεται. Και τώρα που η περιπλοκότητα και το κόστος του Brexit κατέστησαν σαφή, πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε για τη χώρα μας. Είναι ε, απόλυτα απολωμένο και σε αδιέξοδο το Westminster. Πρέπει ο λόγος να επανέλθει στο Βρετανικό λαό. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά, Γκονθάλεφ Πόντ. Αγαπητοί συνάδελφοι, χθε ε, είχαμε αυτή την ψηφοφορία που κατέστησε μόνο ένα σαφέ. Ότι η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε τη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρει τι θέλει. Είχαμε πλειοψηφίε σε δύο αρνητικέ πλειοψηφίε, αλλά καμία πλειοψηφία για τη θετική ψήφο. Μετά από μήνε ε, αυταπατών και ψευδεστήσεων, θα πρέπει επιτέλου το Βρετανικό Κοινοβούλιο να αποδειχθεί την αλήθεια. Το Brexit δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι βρετανικό πρόβλημα. Οπότε σας παρακαλώ βρείτε λύση. Όλοι θέλουν ε, την καλύτερη δυνατή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι το θέλουμε. Αλλά όχι πάση θυσία. Είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να αναμένει από εμά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι να ε, καταρρύψουμε τις αρχές μας. Για έναν απλό λόγο. Το να είναι κανείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οικονομική λύση είναι μια επιλογή ζωή. Είμαστε μια κοινότητα κοινών αξιών που βασίζονται στο κράτο δικαίου και συνθήκε. Δεν είναι απλώ εμπορική σχέση. Η Βρετανική κυβέρνηση δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Η Βρετανική κυβέρνηση πρέπει να το λύσει. Εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε τεθειμένοι να υπογράψουμε οποιαδήποτε συμφωνία αν έλθει σε εμά. Αλλά είμαστε και διατεθειμένοι να συνεχίσουμε χωρί συμφωνία. Μέχρι χθε θεωρούσαμε ότι το Brexit ήταν αντίδραση σε μια ευρωπαϊκή κρίση. Τώρα ξέρουμε ότι είναι αντίδραση σε μια εθνική βρετανική κρίση. Χθε κατέστη σαφέ ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για Brexit με συμφωνία και δεν υπάρχει συμφωνία για Brexit χωρίς συμφωνία. Άρα το πιο λογικό θα ήταν να ηρεμήσετε και να συνεχίσετε να προσπαθείτε. Και στον κύριο Φαράτζ δεν είναι εδώ βέβαια, με κάθε σεβασμό, σας παρακαλώ, να είστε πολύ προσεκτικός όταν χρησιμοποιείτε τη λέξη πόλεμος. Γιατί ναι, υπήρξε πόλεμος και δόξα τω Θεώ τον κέρδισαν οι Βρετανοί. Όλοι πήραμε το ε, μάθημα, αλλά ίσως όχι ο κύριος Φαράτζ. Κύριε Γκονθάλεφ Πόντς, έχετε μια μπλε κάρτα. Από τον κύριο Έθεριτζ. Θέλετε να απαντήσετε. Φυσικά όχι. Είπατε όχι. Ω, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Θα πάω στον Οριλά. Ο κύριος Γκονθάλεφ ε, είπε όχι. Ευχαριστώ. Και τώρα... Φεύγετε κύριε Έθεριτζ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, για δύο λεπτά, η κυρία Ντελάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να πω ότι αυτό που συνέβη χτες ε, στο, ε, στη Βουλή των ε, Κοινοτήτων ήταν κάτι το ιστορικό, κάτι που το περιμέναμε. Βεβαίως, ε, συλλογικά δεν ξέρουν τι θέλουν, μόνο ξέρουν να βγάζουν μεγάλους λόγους κάπως όπως ο κύριος Φαράζ, ο οποίος ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση μια μισή ώρα για το Brexit. Το Brexit είναι raison d'être, δεν μπορεί να παραμείνει ε, σε αυτήν την αίθουσα. Ε, νομίζω ε, μας μίλησε, ήταν στο YouTube και έφυγε. Δεν ξέρει ο κύριος Φαράζ τι θέλει. Αυτό που θέλει είναι το πιο σκληρό Brexit με χωρίς συμφωνία, no deal, για να ε, μπορέσει ε, να καταστρέψει τις δουλειές ε, των συνήθων ανθρώπων και να δημιουργήσει κάτι άλλο. Ακούγοντας τη συζήτηση εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που ακούω από τους συναδέλφους είναι Α καθίσουμε και ας δούμε τι μπορούμε να συμφωνήσουμε για να υπάρξει μια ψηφία και μια λύση. Ε, κάποιος λέει θα προτιμούσε μια τελωνιακή ένωση. Γιατί κανείς δεν προτείνει στη Βουλή των Κοινοτήτων μια τροπολογία γι' αυτό και να δει μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Μια τελωνιακή ένωση θα ήταν η καλύτερη ένωση για να αποχωρήσουν οι Βρετανοί για να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίες από τις δύο πλευρές της μάχη και να βρεθεί μια λύση. Ε, ασχολούμαστε ε, με πολιτική εδώ και στο Westminster όχι μόνο για να βγάζουμε λόγους αλλά για να δημιουργούμε πλειοψηφίες και να βρίσκουμε λύσεις. Ας αρχίσουμε να εργαζόμαστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στη διαδικασία προσοχή του Προέδρου. Αν σεβαστεί το χρόνο, θα ε, μιλήσω στον are περισσότερο. Κύριο Χίρτσο. Political... Οι Βρετανοί φίλοι μα βρίσκονται σε κατάσταση πολιτική σύγχυση σε σχέση με τον Brexit. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε με δημιουργικό τρόπο. Πρώτον, θα πρέπει να, προσθέσουμε, να δώσουμε στου Βρετανού περισσότερο χρόνο για να αποφασίσουν. Δεύτερον, που αποφασίσουν κατά ε, του σκληρού Brexit, τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν και στην ενιαία αγορά ε, και στην Τελωνιακή Ένωση φυσικά. Να δείξουμε ποια ήταν τα σοβαρά λάθη που έγιναν μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματικά ανάγκη το Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε μέρα μας δείχνει ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Αουιλάρα. Πρόεδρε, μια αρνητική πλειοψηφία από ετερόκλητους βουλευτές στην ουσία οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια μακρά και σκοτεινή σύραγγα σύγχυσης και δημιουργούνται προβλήματα σε επίπεδο πολιτικό, σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο γενεών θα έλεγα και διαφορών μεταξύ τους. Η Βρετανική κυβέρνηση οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα το οποίο δυστυχώς δεν έδωσε αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Υπάρχουν εκατομμύρια Βρετανών οι οποίοι άκουσαν με πάρα πολύ υπομονή τα ψέματα και τις ύποπτες δηλώσεις των εθνικιστών και των λαϊκιστών. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα μήνυμα σαφές κατανοητό το οποίο να παρέχει ασφάλεια και εγγυήσεις. Πρέπει να σεβαστούμε τους πολίτες και να τους ελαφρύνουμε από τις επιπτώσεις της ανασφάλειας και της, του φόβου. Κύριο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κρίση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε εδώ. Μιλάμε για τον πλουραλισμό και τον διάλογο και κάθε φορά οι συνάδελφοι που ζητούν τον λόγο τους λένε όχι ε, και όταν θέλουν να θέσουν ένα ερώτημα δεν δέχεται ο άλλος το ερώτημα. Η Ευρώπη μας παρακολουθεί. Η κρίση την οποία ζούμε υπάρχει σε όλες τις χώρες. Υπάρχει και στη Γερμανία. Η στήριξη των δύο μεγάλων κομμάτων έχει μειωθεί. και παρά έναν πρόεδρο ο οποίος στη Γαλλία τον θαυμάζει όλη η Ευρώπη δεν τον θαυμάζουν οι πολίτες του. Αν πράγματι θέλουμε να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή συνεργασία, αν πράγματι θέλουμε η Ευρώπη να συνεχίσει να υπάρχει, θα πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές μας, γιατί η πολιτική μας απειλεί και απειλήσε τους Βρετανούς. Μετανάστευση, ευρωπαϊκό στρατός, κοινό νόμισμα, αν τα αλλάξουμε όλα αυτά τότε θα αλλάξουμε σωστά την Ευρώπη. Ο κύριος Χατζηγεωργίου για ένα λεπτό. Έχει δώσει κατεύθυνση προς το Βουλή των Κοινοτήτων για επαναπροβληματισμό και νομίζω ότι και εγώ γενικά πράγματα μπορεί να πω. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ψες δεν ήταν ήττα της Βρετανικής κυβέρνησης μόνον ήταν ήττα κατά την άποψή μου της μεγαλαυχίας των πολιτικών εξουσιών διαχρονικά και βεβαίως της βρετανικής μεγαλαυχίας διαχρονικά. δεύτερο πρέπει να κάνουμε αναφορά σήμερα σε ένα όνομα ένα ένεκεν του οποίου βρισκόμαστε σήμερα εδώ και ένα και του οποίου βρίσκεται ολόκληρη η ευρωπαϊκή ένωση και η βρετανία σε αυτή την κατάσταση και είναι το όνομα του κυρίου David Cameron. Γιατί το λέω, όχι για να χλεβάσω, αλλά για να πω ότι οι μεγάλοι ηγέτες στις κρίσιμες ώρες δεν κάνουν παιχνίδια δεν παίζουμε χαρτοπέγνιο δεν είμαστε γκάμπλερς. το τρίτο δημοψηφίσματα πρέπει να γίνονται με φιδό ιδιαίτερα όταν οι σημερινοί αποφασίζουν για το πώς θα ζουν εδώ οι άνθρωποι έναν αιώνα μετά. με φιδό τα δημοψηφίσματα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλά αρνητικά πράγματα συμβαίνουν. Αυτό είναι άσχημο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Συμφωνώ. Οι, οι Βρετανοί εκλογής ε, παρεπλανήθησαν μέσω ψεμάτων. Τώρα πληρώνουμε το τίμημα στον λαϊκισμό. Τώρα ε, γνωρίζουμε τι σημαίνει μία συμφωνία. Τι έχουμε ενώπιον μας. Ε, ή να αποχωρήσουν χωρίς συμφωνία ή παραμονή. Να αποφασίσει ο λαός. Πολλές επιχειρήσεις εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Και πολλοί Βρετανοί πολίτες ζητούν ε, υπηκότητα άλλης χώρας της Ένωσης. Εγώ είμαι υπέρ περισσότερης Ευρώπης. Ήθελα να απαντήσω στον κύριο Καμάλ, επικεφαλή των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και στον κύριο Φάρατζα, αλλά έφυγαν. και οι δύο. Βεβαίω. δεν του ενδιαφέρει η συζήτηση, μόνο να μιλήσουν. Ο Ντέιβιτ Κάμερον έχει την ευθύνη του Brexit, διότι ζήτησε ε, από το λαό να ψηφίσει, ήθελε να επεκληγεί βεβαίω. Θα ήθελα να χαιρετήσω, να συγχαρώ τον Μισελ Μπαρνιέ και την ομάδα του, διότι δικαίω λέει ότι αυτή η συμφωνία των 600 σελίδων είναι ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Και βεβαίω το πρόβλημα θα παραφράσω την ε, Μάργαρετ Θράτσερ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση η μόνη εναλλακτική είναι η χαοτική ε, κατάσταση σήμερα. Θα μπορούσε να δώσει χρόνο στο χρόνο και στο επίπεδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι πέραν από τους λαϊκιστές ε, είναι η λογική ε, που θα υπερισχύσουν διότι έχουμε όλοι συμφέρον να παραμείνει. Δεν θα υπάρξει Brexit. Το κύριο Στάμπατ. Κυρία Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι απέτυχε η συμφωνία που ήταν επιτάπητος. Οπότε ή θα υπάρξει ένα καταστροφικό Brexit που θα δημιουργήσει προβλήματα και στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε το μόνο που μένει είναι να ρωτήσουμε το λαό. Αλλά βεβαίω ορισμένοι λένε, μα του ρωτήσαμε ήδη. Δεν είναι δημοκρατικό να του ξαναρωτήσουμε. Αλλά η δημοκρατία, η δημοκρατία είναι η κυριαρχία του λαού και δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε ένα λάθο. Το καλύτερο θα ήταν να ξαναρωτηθεί ο λαό. Με το ερώτημα. Θέλετε σε διαπραγματεύσει με τα θεσμικά όργανα να βρείτε μια άλλη λύση. Και θέλω να κάνω πραγματικά παράκληση προς το σώμα αυτό. Δεν πρέπει να διαπραγματευόμεθα υπεροπτικά. Όλα όσα άκουσα εδώ ε, είναι να τιμωρηθεί η Βρετανία. Αυτή είναι η λάθος προσέγγιση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ευρώπη. Εάν γίνει έτσι συζήτηση θα καταλήξουμε θετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάνναγκαν, επόμενο. Το πρώτο που πρέπει να υποθεί και δεν, συμφωνεί, δεν συμφωνώ συχνά με τον Κέλλη είναι να επανέλθουμε σε αυτό που είπε η Αλίν Φώστα ότι δεν πρέπει να υπάρξουν ποτέ σκληρά σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν υπήρξαν ποτέ σκληρά σύνορα. Μα πού ήταν όταν υπήρξαν ε, σκληρά σύνορα. Ίσως για εκείνη δεν, ε, δεν ε, υπήρχαν για εκείνη, αλλά είχαμε σκληρά σύνορα. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε παράταση του άρθρου 50. Αυτό το σκάκι που παίζεται δεν θα καταλήξει καλά. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μας εξηγήσει πώς θα βοηθήσει την Ιρλανδική οικονομία και ιδιαίτερα τους γεωργούς μας. Άκουσα ε, ένα σχόλιο από τον Κονθάλεθ Πόντ ότι δεν είναι πρόβλημα τη Ευρώπη. Αλλά βεβαίω, ναι, δεν το δημιούργησε η Ευρώπη και αυτό το κατανοώ. Βεβαίω αλλά όσο και να το πούμε, είναι τώρα, έχει καταστεί και δικό μα πρόβλημα. Εμεί στην Δημοκρατία τη Ιρλανδία είμαστε μέλο τη Ένωση. Μα δημιουργεί τρομερά προβλήματα η κατάσταση. Το να λέτε ότι δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα λοιπόν είναι λάθο. Πρέπει να αλλάξετε στάση. Και κύριε Μπαρνιέ, Πρέπει να πω ότι ανησυχούσα στην αρχή για σας, αλλά έκανε καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια, κρατήσατε την ψυχραιμία σας όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φράγκαλη, πρόεδρος. Ε, τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Χόκμαρκ. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα σχετικά με τους συναδέλφους του UKIP από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν ούτε μία έδρα στο Westminster. Καμία έδρα εκλεγμένη από τον λαό της Μεγάλης Βρετανίας για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Και νομίζω ότι έχει σημασία αυτό. Αλλά επίσης ο κύριος θα ήσασταν ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχατε καμία αντιπροσώπευση κοινοβουλευτική, πουθενά. Δεύτερο, σχετικά με τους Βρετανούς φίλους μας και με αυτούς που ασχολούνται με το θέμα στο Westminster. Αν θέλουν παράταση, χρόνο για προβληματισμό, αν θέλουν να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελαμε να τους πούμε ότι είναι πρόσδεκτοι. Και η κυρία Γραπίνη τώρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Πάρα πολλά πράγματα λέχθηκαν εδώ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ε, σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει μεταξύ μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διαπραγματευτή. Το πρόβλημα δεν δικό μα, αλλά είναι πρόβλημα τη μεγάλη Βρετανία. Ε, και θέλω ε, να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον των πολιτών μα που ζουν εκεί και αυτών τη μεγάλη Βρετανία που ζουν εδώ. Το μέλλον το εμπορικό, όχι μόνο πρέπει να συνεχίσουμε τη τη διαπραγμάτευση, αλλά θα πρέπει και ο πληθυσμό ο οποίο στην πλειοψηφία του θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγα στο Λονδίνο, στο Μπέρμιγκα, μίλησα με τους πολίτε με τους επιχειρηματίε. Θέλουν ε, να παραμείνουν. Είναι οι πολιτικοί άνδρες που δίνουν την κατεύθυνση αυτή της δεξιάς που ε, ρίχνουν μηνύματα που λένε ότι αν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα πληρώνουμε εμείς ε, τις συντάξεις στους Μεγάλους Βρετανούς. Ωραία, τώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία κάτω του και δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμαντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς την συμπαράσταση των Βρετανών στην πιο δυσχερή και πιο ζωφερή στιγμή της ιστορίας μας δεν θα ήμασταν εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Και η δική μου χώρα ε, είναι ευγνώμων για την ελευθερία που μα έδωσαν οι Βρετανοί στρατιώτε. Είναι άρρηκτη η δεσμή μεταξύ τη Βρετανία και τη Ευρώπη, Είτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Πάντα θα είναι τμήμα τη Ευρώπη η Βρετανία. Με έναν τρόπο που θα καθορίζει το κοινό μα πεπρωμένο. Και λυπάμαι που βλέπω να είναι τόσο διηρημένο όσο σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαιρέσει που έχουν, που έχουν προκληθεί από τον Brexit έχουν παραλύσει την Βρετανική κοινωνία. Εγώ θα παραμείνω αιώνια ευγνώμων. Όχι μόνο για την ελευθερία μας, αλλά και για τους Βρετανούς ε, δασκάλους που είχα όταν ήμουν νέος, που μου έμαθαν να αγαπώ τη Βρετανική λογοτεχνία, την τέχνη, μου έμαθαν τη γλώσσα. Αυτό δεν θα αλλάξει, ό,τι και να συμβεί. Αλλά θέλω να καταστήσω κάτι απόλυτα σαφές, αντιδρώντας ορισμένα που ελέγχθησαν από τον κύριο Καμάλ και τον κύριο Φαράτζ. Εγώ στην Επιτροπή με τον Μισελ ούτε σε καμία από τις 27 πρωτεύουσες δεν διαπίστωσα καμία τιμωρητική διάθεση σε αυτή τη διαδικασία. Κανείς δεν θέλει να τιμωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο που αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις διαπραγματεύσεις σε όλες τις πρωτεύουσες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η στάση μας ήταν να γίνει η μικρότερη δυνατή βλάβη σε αυτή τη διαδικασία αλλά να μην αυταπατώμεθα ζημιά θα γίνει. Το Brexit θα κάνει ζημιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η κοινή μας ευθύνη να περιορίσουμε αυτή τη βλάβη όσο γίνεται. Τι θα γίνει τώρα στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια. αυτό θα το αποφασίσει ο Βρετανικός λαός. Και πρώτα απ' όλα η Βουλή των Κοινοτήτων, όπου θα γίνουν οι συζητήσεις. Εμείς ε, θα παίξουμε το παιχνίδι όπως θα καθορίσει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο πώς θα παιχθεί περαιτέρω. Ε, ποτέ δεν έκρυψα. Θα προτιμούσα να παραμείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό εξαρτάται από τους Βρετανούς πολιτικούς, όχι από εμά. Και κάτι που θέλω επίσης να καταστήσω σαφές, επειδή άκουσα τον κύριο Καμάλ που είπε ότι υπάρχει ενιαία αγορά και άλλα στοιχεία. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει θα φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα κρατήσω όλα τα στοιχεία που μου αρέσουν χωρί να καταλαβαίνει πώ θίγει αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ω Ευρωπαίοι πολιτικοί, ω κράτη-μέλη, ω θεσμοί, έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε το ουσιώδη στοιχεία του τι σημαίνει να είναι κανεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το αδιέρετο των τεσσάρων ελευθεριών. Είναι η ακαιρεότητα τη ενιαία αγορά. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάτι που με καταπλήσει επίσης είναι ότι ο κύριος Φάρατζ έχει αυτό το όνειρο, το ψευδές όνειρο περί ανεξαρτησίας, που τον οδηγεί στο να αγνοεί εντελώς τη θεμελιώδη σημασία της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής για την ειρήνη στην Ευρώπη. Είναι απόλυτα σαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουμε συλλογική ευθύνη ως Ευρωπαίοι να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η ειρήνη στο νησί της Ιρλανδίας. Και με βάση την ανάλυση μας για να υπάρξει αυτή η ειρήνη δεν πρέπει να υπάρχουν σκληρά σύνορα στο νησί της Ιρλανδίας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τον backstop. Και αυτό είναι διαπραγματευτό. Και πραγματικά τρελαίνεται ο άνθρωπος όταν ε, από τη μία βλέπει να υπάρχει τέτοια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που κανείς στις 27 ε, ε, πρωτεύουσε λέει ε, δεν θεωρεί ότι μπορούμε να εγκαταλείψουμε την Ιρλανδία. Και πολλοί στο Westminster δεν βλέπουν την ουσιώδη αξία τη Συμφωνίας Μεγάλης Παρασκευής. Και γι' αυτό το όνειρο της υποτιθέμενης εξαρτησίας είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την ειρήνη στην Ιρλανδία. Και δεν μιλάω για τις δουλειές, τις επενδύσεις και όλα αυτά θα ήταν ειλικρινές. Σε αυτή την εκστρατεία που οδήγησε στην ε, απόφαση για τον Brexit, την οποία απόφαση σεβόμεθα. Θα ήταν καλό να πούνε ότι θέλουμε τόσο πολύ την ε, ελευθερία μας που δεν, θέλουμε, που δεν μας ενδιαφέρει αν θα χάσετε δουλειά για τις επενδύσεις, για το σύστημα υγείας. Δεν μας ενδιαφέρει ότι θα υπάρχουν ποτηγιαρίσματα στους δρόμους. Θέλουμε την ανεξαρτησία μας ανεξαρτήτως συνεπειών. Αυτό θα ήταν μια ειλικρινής προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Brexit. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στο Westminster, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε ειλικρινά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει όσο λιγότερο μικρότερη ζημιά, όπως και αν διαμορφωθεί η κατάσταση. Κύριε Καμάλ, αναφερθήκατε στους Eagles. Εγώ θα αναφερθώ στους Rolling Stones. Δεν μπορείς πάντα να ε, αποκτήσεις αυτό που θέλεις, αλλά αν προσπαθήσεις αρκετά σκληρά μπορεί να αποκτήσεις αυτό που χρειάζεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βεβαίως ε, ε, θα θέλαμε όλοι εδώ να έχουν την ίδια απόψη και τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Τσιότ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι θα πρέπει να ελπίζουμε ότι οι βουλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα οδηγήσει ε, σε συντεταγμένη έξοδο και θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια τέτοια διαδικασία. Εάν αυτό το θετικό σενάριο υλοποιηθεί, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η συμφωνία της 25ης Νοεμβρίου ήταν το πρώτο βήμα σε μια μακρά διαδικασία. Θα πρέπει η εφαρμογή ε, του συμφωνίας αποχώρησης να παρακολουθείτε στενά, ούτως ώστε να έχουμε αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών επιχειρήσεων και οι διαπραγματεύσεις των μελλοντικών σχέσεων να οδηγήσουν σε αυτό. Θα πρέπει να βασιζόμαστε στη συνεργασία σας σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ άλλη μία φορά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Έκλεισε η συζήτηση. Ευχαριστώ. buenos Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσετε μαζί μας, να συζητήσετε με τους Ευρωπαίους βουλευτές για την θέση της Ισπανίας στην Ευρώπη. Σήμερα είναι μια μέρα πολιτικά πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε πάντα ανοιχτό το θέμα του Brexit αλλά είναι σημαντικό για μας να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν σημασία, το θέμα της μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει και έχει ψηφίσει την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Περιμένουμε τώρα τις χώρες μέλη και το Συμβουλίο να υπερψηφίσουν και τη δική μας πρόταση έτσι ώστε να καταλήξει μια διαδικασία και μια συζήτηση γύρω από τα θέματα ε, των προσφύγων και της ε, μετακίνησής τους και της μετεγκατάστασής τους. Εμείς ζητάμε να περάσουμε από το 1,1 στο 1,3 του προϋπολογισμού για τους πόρους της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα δημιουργήσει θέματα στα κράτη-μέλη, αλλά με τους ιδίους πόρους θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις διαφορές αυτές και εδώ η συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή. Υπάρχει μια πρόταση λοιπόν από πλευρά στο Κοινοβουλίου και αυτό που έχει σημασία για μας είναι να υπερασπιστούμε την θέση μας μια θέση κεντρική, μια θέση καρδιά της ευρωπαϊκής εξέλιξης Φυσικά έχουν περάσει τώρα και αρκετά χρόνια μετά από την ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να χαιρετήσει και τον κύριο Μπορέλ, τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας που ήταν πρόεδρος αυτήν εδώ την αίθουσα. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ και σας δίνω αμέσως το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι τιμή, πραγματική τιμή η δυνατότητα που μου δίνετε να περθώ σε εσά για να σας μιλήσω για την ε, θέση της Ισπανίας σε αυτή την ε, συναρπαστική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και είμαι πεπισμένος ότι είναι συναρπαστική και με βάση τη δική μου εμπειρία το 1985 όταν υπεγράφει η ένταξη Τη Ισπανία στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ε, ήμουν 13 ετών. Και παρά το ότι πέρασε τόσο χρόνο, θυμάμαι πολύ σαφώ εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι τη συγκίνηση που αισθανθήκαμε εμεί που κατά δεκαετίε ε, υποφέραμε λόγω έλλειψη τη δημοκρατία και των ελευθεριών στην Ισπανία. Θυμάμαι τη συγκίνηση μια γενιά, ε, ολόκληρη Ισπανών, τη γενιά των γονέων μου, ανδρών και γυναικών, για του οποίου η Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια τη δικτατορία, σήμαινε ελευθερία, κράτος δικαίου, συνοχή και πρόοδος. Εκείνη τη στιγμή ε, εκπροσωπούσε πολλά για την Ισπανία. Ιδιαίτερα την εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει πισωγύρισμα. Ότι επιτέλους ήμασταν σε ειρήνη με την ιστορία μας. Ότι επιτέλους κανείς ποτέ δεν θα μας ε, αφαιρούσε τη δημοκρατία πλέον. Έκτοτε, οι επόμενες γενιές ε, Ισπανών, όπως η δική μου, είδαν τα εσωτερικά σύνορα να γίνονται ανάμνηση της ιστορίας και είδαν ε, να υπάρξει ότι υπάρχει αλληλεγγύη και σχέση με λαούς που παλιά ήταν μακρινοί. Πάντα ε, σε σεβασμό με τις αξίες που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές, η νομική ε, ασφάλεια, ο διάλογος, η αποδοχή των άλλων, ο φεμινισμός, η ισότητα ευκαιριών, η αδελφότητα, η συνύπαρξη, η οικολογία και η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών. Οπότε, βεβαίως, είμαι ένθερμος Ευρωπαίος. Είμαι περήφανος για τι εκπροσωπεί αυτό. Και ιδιαίτερα περήφανος τώρα που ορισμένοι προβάλλουν τον αντιευρωπαϊσμό για να επιτύχουν εκλογικά ωφέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε Ταγιάννη που μου δίνει την ευκαιρία να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο που είναι στην καρδιά αυτής της συζήτηση, που είναι μια μεγάλη πρόκληση. Τώρα που πρόκειται να εορτάσουμε την 40η επέτειο των πρώτων άμεσων ευρωπαϊκών εκλογών. Η Ένωση βασίζεται στην προτεραιότητα των δημοκρατικών αρχών. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, πριν απ' όλα, θα ήθελα να αναφέρω την ψηφοφορία που έγινε χθε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Σέβομαι, αλλά σέβομαι ως ε, πρόεδρος της κυβέρνησης ενός κράτους μέλους, αλλά λυπάμαι επίσης για την ε, απόρριψη της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια συμφωνία την οποία διαπραγματευθήκαμε για πάνω από 1,5 χρόνο. Και θέλω να αποδίσω φόρο τιμής στον ε, Μισελ Μπανιέ. Έκανε καταπληκτική εργασία για να διατηρήσει την ενότητα των 27 κρατών μελών. Όπως έλεγα, αυτή η συμφωνία ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευση για 1,5 χρόνο και νομίζω ότι είναι η καλύτερη εφικτή συμφωνία. Είναι η λύση που προστατεύει καλύτερα τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και του συνόλου των κρατών μελών τη Ένωση. Άρα τη Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Είναι η λύση που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών αλλά και τα δικαιώματα των ε, επιχειρήσεων. Είναι μια συμφωνία που έχει παραχωρήσει και από τι δύο πλευρέ. Είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει κανεί κάτι τέτοιο, μια ισορροπία που επιδιώκει πρώτα απ' όλα μια συντεταγμένη έξοδο. Ε, άρα τώρα είναι θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκρίνει τι αποφάσει που θεωρεί κατάλληλε για τα επόμενα βήματα. Εμεί, ω κράτη-μέλη και ω ε, ενωσιακοί θεσμοί, κάνουμε τη δουλειά μα. Και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνουμε τα αναγκαία μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε την επίπτωση μιας ενδεχόμενη άτακτη αποχώρησης. Κυρίε και κύριοι, πάντα εξέφρασα τη γνώμη μου και στο Ισπανικό Κοινοβούλιο αλλά και στις διάφορες ε, συνεντεύξει που έχω δώσει πάντοτε έχω τονίσει ότι είναι λάθος το Brexit και για την ε, Μεγάλη Βρετανία και για την Ένωση. Όλοι χάνουμε. Και ιδιαίτερα η Βρετανία όμω. Ιδιαίτερα εκείνοι που χρειάζονται περισσότερο την προστασία τη κυβέρνησή του. Δηλαδή οι πιο ευάλωτοι. Αλλά είναι μια κυρίαρχη απόφαση την οποία ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σεβαστούμε. Γι' αυτό επιθυμώ το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει την πιο στενή σχέση με το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση όμω είναι δική του. Αλλά οι αρχέ μα είναι σαφεί. Η ε, ακαιρεότητα τη εσωτερική αγορά, ε, το αδιέρετο των τεσσάρων ελευθεριών, και η αυτόνομη λήψη αποφάσεων από την Ένωση. Στα πλαίσια αυτών των τριών σημείων πάντα θα παραμείνουμε. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα μιλήσω για την ε, ανάγκη να κινητοποιηθεί η Ευρώπη. Για την ανάγκη να αποκτήσει νέα νομιμοποίηση η Ευρώπη ε, έναντι των νέων ε, προκλήσεων. Αλλά και έναντι εκείνων που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη. Υπάρχουν διάφοροι εντό και εκτό σημαντικοί παράγοντε που θέλουν να καταστραφεί η Ένωση. Ω επικεφαλή Ω συγγνώμη, όπω ω ηγέτη τη σοσιαλδημοκρατική οικογένεια, βεβαίω ε, θα περιμένετε να μιλήσω για την ε, κοινωνική Ευρώπη, για την Ευρώπη που προστατεύει. Και θα το κάνω, γιατί η, Ευρώπη, η κοινωνική Ευρώπη είναι η Ευρώπη των πεπιθήσεων. Και για αυτόν τον λόγο, για αυτή την ε, ηθική πεποίθηση, γιατί θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη αυτό που αναμένουν οι πολίτε από αυτήν, διαρωτάμε ποια είναι η κεντρική ιδέα τη ομιλία μου. Θα είναι κάτι πολύ πιο απλό. Το συνοψίζω σε μια φρόση. Η Ευρώπη για να μπορεί η Ευρώπη να προστατεύει, σε αυτή την ιστορική συγκυρία πρέπει εμεί να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε μια Ευρώπη ε, ε, δικαιωμάτων που να προστατεύει του πιο ευάλωτου. Να προωθήσουμε μια Ευρώπη που να δίνει ευκαιρίε για του νέου μα και για του ε, μακροχρόνια άνεργου. Σε χώρε όπω η δική μου, οι μακροχρόνια άνεργοι δεν είναι μόνο 60 ετών, μπορεί να είναι και 45. Και πάσχουν από την Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη που να ενισχύει τον κοινωνικό ιστό αλλά και τον ε, ε, επιχειρηματικό ιστό και να προστατεύει εκείνους που πάσχουν από την επισφάλεια. Πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την ε, άμυνα των συμπολιτών μας ούτω ώστε η Ευρώπη να γίνει ένα παγκόσμιο παράγοντα που να μπορεί να σεβαστεί τι αξίε και τα ιδανικά του. Η προστασία τη Ευρώπη είναι να τονίσουμε ότι πιστεύουμε στη Συμφωνία των Παρισίων για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε μια για πάντα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μόνο έτσι, με μια Ευρώπη που να ε, με του πολίτε τη. Μια αυτόνομη Ευρώπη που να υπερασπίζεται το κοινωνικό τη μοντέλο. Μια Ευρώπη που θα ολοκληρώσει την οικονομική και νομισματική τη ε, δομή. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει που θα έχουμε την ε, επόμενη δεκαετία με επαρκή εγγύησεις. Τι επόμενες δεκαετίες. Δεν πρέπει λοιπόν να αμφιβάλλουμε. Στους εχθρούς τη Ευρώπη πρέπει να του πω η πεποίθησή μας και η αποφασιστικότητά μας θα νικήσουν την, ε, τον αυταρχισμό. Ορισμένοι έχουν μια ρητορική που αποκλείει άλλους. Ορισμένοι έχουν ε, πολλοί με μεθόδου και λένε ψέματα. Είναι η στιγμή εμεί να αποδείξουμε την πεποίθησή μα, την αποφασιστικότητά μα για να υπερασπίσουμε το κοινό μα εγχείρημα που είναι η Ευρώπη. Σήμερα γίνεται μια πραγματική μάχη ε, ιδεών. Αυτό είναι ένα πλαίσιο ε, που έχουμε σε όλε μα τι χώρε και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, πρέπει να υπάρξει οπισθοχώρηση ή πρόοδο. Εμεί θέλουμε το, να είναι σαφέ ότι το μέλλον ποτέ δεν κατακτήθηκε με υποχωρήσει. Γι' αυτό δεν θα κάνουμε καμία υποχώρηση στην ε, υποστήριξη του ευρωπαϊκού μοντέλου. Η Ευρώπη προστατεύει του πάντε. Όλοι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, όχι μόνο η κοινωνία των πολιτών. Το σύνολο τη κοινωνία πρέπει να προστατεύσει την Ευρώπη. Σε αυτού που στέλνουν μηνύματα εσωστρέφεια, ε, ακόμη και από εδώ, η Ευρώπη για μένα δεν είναι ούτε ποτέ θα είναι απειλή στην καταπληκτική πολυμορφία των χωρών μας, των γλωσσών μας και των πολιτισμών μας. Η Ευρώπη είναι ακριβώς το αντίθετο. Η Ευρώπη ε, αυξάνει, πολλαπλασιάζει, δεν διαιρεί τις ταυτότητες. Αν είσαι Ευρωπαίος δεν είσαι λιγότερο πάνω το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι απλώς μια γεωγραφική έκφραση. Ήταν και είναι κοινότητα αξιών. Των αξιών της ε, Γαλλικής ε, Επανάστασης, ελευθερία, ισότητα και η αδερφότητα που είναι τόσο σημαντική σήμερα. Αυτέ είναι οι αξίε ανοιχτών κοινωνιών, αισιοδόξων κοινωνιών που καινοτομούν, που δημιουργούν, που θεωρούν ότι το μέλλον είναι ευκαιρία, ποτέ απειλή. Είναι κοινωνίε που συνδέουν την αναγκαία ανταγωνιστικότητα για την οικονομική ανάπτυξη με κάτι που είναι θεμελιώδε, που μα καθορίζει ως Ευρωπαίου, που είναι η κοινωνική συνοχή και το μοντέλο μα ευημερία. Αυτή η δεσμευσή μα που μα ενώνει Όπω για παράδειγμα οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη ε, του θεματολογίου 2030 που είναι ένα πραγματικό συμβόλαιο τη επόμενη δεκαετία που θα κάνει την Ευρώπη τον κύριο ε, πρωταγωνιστή αυτή τη προσπάθεια. Είναι προφανέ ότι υπάρχει κοινωνική απογοητεύση στα πλαίσια τη παγκοσμιοποίησης. Το βλέπουμε στις ε, πόλεις μας, στους δρόμους μας, στι πλατείε μα. Αυτή η απογοήτευση ευνοεί βεβαίως τη ρητορική των ακραίων έχουμε μια τεράστια, ένα τεράστιο παράδοξο. Πρώτα απ' όλα η παγκοσμιοποίηση ανακατένει με την, τον πλούτο μεταξύ περιοχών του κόσμου, άρα μείωσε την παγκόσμια ανισότητα, αλλά αυξάνει την ανισότητα, αυξάνει συγγνώμη, την, την ανισότητα στο εσωτερικό των κοινωνιών μα. Και αν το σκεφτούμε καλά, η αύξηση του αντιευρωπαϊσμού οφείλει πολλά σε αυτό το τελευταίο φαινόμενο. Αλλά η παγκοσμιοποίηση δεν είναι θεομηνία που μας βρίσκει ανυπεράσπιστους. Ο Γκέτα έλεγε ότι τα... οι γονεί θα πρέπει να δουν στα παιδιά του ρίζε και φτερά. Παρόμοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει στου πολίτε τη ρίζε, δηλαδή μια βάση στήριξη, μια προστασία, αλλά και φτερά. Δηλαδή να τους δώσει δυνατότητες για να, είναι, ε, ε, να έχουν ευμάρεια και να έχουν δυνατότητες σε έναν παγκοσμιμένο... Ε, είμαστε σε μια κοσμοστορική αλλαγή. Στι 26 Μαου θα ανοίξει ένα νέο κύκλο πολιτικό για την Ευρώπη. Και θα πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν την παγκοσμιοποίηση για να εξακολουθήσει να ισχύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Θα πρέπει να εδραιώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση συμπληρώνοντά την με την αναγκαία πολιτική, κοινωνική και θέλω να να